ανακοίνωση όσον αφορά την εκλογή των αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου. Προτείνω ε, να πούμε ότι σήμερα μέχρι τις 22 και 30, μέχρι τις 10 και 30 ε, να υπάρχει προθεσμία υποβολής των ε, υποψηφιωτήτων για, την, για τις θέσεις των αντιπροέδρων και θα πρέπει να υποβληθούν στην αίθουσα R00100.